καλωσορίζω όλους τους βουλευτές. Έχω ανακοίνωση να σας κάνω. Στις 16 Ιουλίου του 2009 υπέβαλα στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων μία ε, αίτηση άρση ασυλίας ενός βουλευτού. Το 2010 ο πρόεδρος της Νομικής Επιτροπής με ενημέρωσε ότι δυνάμη του ψηφίσματος του Απριλίου 2009 του Κοινοβουλίου σχετικά με τους κανόνες ασυλίας ε, που ισχύουν στην Πολωνία ε, έκρινε η Νομική Επιτροπή ότι έτσι αυτή ήταν απαράδεκτη. Άλλο θέμα στην ημερήσια